Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε. Να αρχίσουμε το πρωινό εργασίες Με τις ψηφοφορίες. Πρώτα θα ψηφίσουμε την έκθεση Νταντά για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού. Όπως θα θυμάστε, στις συνεδρίες 14 Η Ιουλίου αποφασίσαμε να ζητήσουμε άδεια να συντάξουμε έκθεση, ε, γνωμοδότηση με βάση το άρθρο 53 του Σωτερικού κανονισμού ε, επί της εκθέσεως πρωτοβουλίας της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού». Η, ε, την γνωμοδότηση την ανέλαβε το ΕΛΚ και η ορίστηκε ο κύριος Δαντά. Στι 30 Αυγούστου είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε και το σχέδιο γνωμοδότηση υπευλήθη στις 12 Οκτωβρίου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 18 Οκτωβρίου και κατατέθηκαν 128 τροπολογίες και 15 συμβιβαστικέ προκειμένου να διευκολυνθεί η σημερινή ψηφοφορία. Ε, αν θέλει ο κύριος Δαντά το λόγο μπορεί να τον λάβει, είδαμε θα ξεκινήσουμε αμέσως την ψηφοφορία της γνωμοδότησής του. Ο συνήθως, τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και τις υπόλοιπες διανατάσσεως της χειρός. Συμβαστική τροπολογία μη, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β, B, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 16, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίψατε. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον. Άρχεται ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, όπως είπαμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 32 τώρα της κυρίας Ροντρίγκε. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 38, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D, ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ή e, ε, ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 του κυρίου Άγνιου. Ποιος είναι υπέρ, διαρατάσεις της χειρός, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 του κ. Μποβέ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Νταντάν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία F, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 τώρα. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 108. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική I. Περνάμε στην τροπολογία 88 του κυρίου Χαΐτεμα. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101 τώρα. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Κ. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία είναι άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε δυνατάσεις της χειρός 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. Τροπολογία 1. Νταντά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3 του κυρίου Νταντάν και πάλι υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α, ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και συγχαρητήρια κύριε Νταντά. Σας δίνω μάλιστα και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το επιτελείο των εισηγητών με το οποίο εκπονήσαμε την έκθεση. Νομίζω ήταν εύκολο τελικά να συμπλήσουμε τις απόψει μα και να καταλήξουμε σε συμφωνία οι πολιτικέ ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το βοηθό μου που πραγματικά ε, με βοήθησε πολύ σε αυτή την έκθεση. Επίσης, ε, ε, τα εύσημα προς τον συνάδελφο Στάζη της ε, κύριας Επιτροπής που συνέταξε την έκθεση πρωτοβουλίας και μάλιστα είχαμε κάπως ε, ιδιόρυθμη ε, κατάσταση γιατί κάπου, προλάβαμε κάπως τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας και κατάφερε να συμπεραλάβει βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης στη δική του έκθεση που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στην αρμόδια κατουσίαν επιτροπή. Τον ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της Επιτροπής μας. Επίση, ε, έχουμε και τα αποτελέσματα της ε, ομάδας εργασίας της Task Force, που είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά της Επιτροπής Γεωργίας. Οπότε στέλνουμε ένα ξεκάθαρο και χειρό μήνυμα προς την Επιτροπή για το έργο που καλείται να πραγματοποιήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Νταντά. Πραγματικά εξαιρετικό το έργο σας. Περάμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης τη δεύτερη ψηφοφορία του πρωινού με την ψηφοφορία της έκθεσης ε, της, του σχεδίου ε, ψηφίσματος που ε, έχει κατατεθεί με βάση το άρθρο 106 παράγραφος 3 που προτείνει τροποποίηση του σχεδίου οδηγίας, της εκτελεστικής οδηγίας των παραρτημάτων 1-5 της οδηγίας 2029 του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και ε, ε, αποτρέπει την εξάπλωσή τους στην κοινότητα. Εμείς θα ψηφίσουμε ένα σχέδιο ψηφίσματο που αντιτίθεται στην εκτελεστική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετική απόφαση την είχαμε λάβει στη συνεδρίαση των συντονιστών τη 8η Νοεμβρίου. Και μάλιστα την ίδια μέρα, λίγο πριν την απόφαση των συντονιστών, είχαμε παρουσίαση τη Γενική Διεύθυνση Άντε και ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας. Ε, μια νέα ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα χθες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, υιοθετήσει την εκτελεστική της οδηγία τον Ιανουάριο, οπότε κρίναμε σκόπιμο να ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος, προκειμένου να έχουμε χρόνο για να καταθέσουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει το Δεκέμβριο είναι φυσικά την τελική απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση της εκτελεστικής οδηγίας προς την οποία αντιτιθέμεθα. Θα ήθελα επίσης να σας εξηγήσω ότι με βάση το άρθρο 106 παράγραφος 3 δεν ε, χρειάζεται πάντα να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακαλέσει την εκτελεστική της οδηγία. Μπορούμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει την εκτελεστική της οδηγία με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχετικές ε, τροπολογίες που προτείνουμε. Και η κυρία Γιλέρα τέτοιε ε, αλλαγέ προτείνει στο σχέδιο εκτελεστικής οδηγία. Έλαβε χώρα η γραπτή διαδικασία μεταξύ των συντονιστών και μάλιστα η πλειοψηφία των συντονιστών τάχθηκε υπέρ της σημερινής ψηφοφορίας του σχέδιου ψηφίσματος. Και είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Γεωργίας ε, καταθέτει αντίρρηση στο σχέδιο μιας εκτελεστικής οδηγίας. Και μάλιστα σήμερα θα ψηφίσουμε. Και μάλιστα άλλες επιτροπές ήδη έχουν εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων. Ζητήθηκαν κάποιες κατατμήματα και ξεχωριστές ψηφοφορίες. Έχουμε ένα νέο κατάλογο ψηφοφορίες. Σας τον έχουμε μοιράσει. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία του σχεδίου ψηφίσματος. Δυστυχώς μερικές ε, προτάσεις για ξεχωριστές ψηφοφορίες ε, υπευλήθησαν ε, πολύ αργά το βράδυ. Θεωρώ ότι καλύτερα είναι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την πρώτη τροπολογία υπαριθμών 2 ξεχωριστά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η τροποποίηση 2. Τροποποίηση 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα και σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα. Voilà. On continue On continue Parfait, on continue, on continue. Donc euh, la Slovénie. Donc... Α συνεχίσουμε την μερίσια διάταξη. Αν μπορείτε να αποχωρείτε με κάποια ε, ησυχία, Μερίσια διάταξη τώρα. Παρουσίαση έκθεση για την αποστολή στη Σλοβενία 21 με 23 Σεπτεμβρίου για την προσωπία της Επιτροπής Γεωργίας και αναπτύξεως της Υπέθρου μετέβη στη Σλοβενία τον μήνα Σεπτέμβριον και είχα την τιμή και το προνόμιο να εγούμε τις γιατί ο κ. Σικέρσκι την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Όλα πήγαν υπέροχα. Η επισκέψη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπόγκοβιτς που ε, διοργάνωσε και με τέριο τρόπο την αποστολή για να αναφερθεί στα αποτελέσματα της επισκέψεως που ενεπλούτησε τις γνώσεις όλων των μελών. Έχετε το λόγο λοιπόν. Λίγη προσοχή παρακαλώ. Ας σεβαστούμε τον ε, ομιλητή. Όσοι πρέπει να καταλήψουν την αίθουσα, ήσουν ε, ήσυχα. Κύριε Μπόγκοβιτς, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ που ηγήθηκατε της ομάδας των μελών της Επιτροπής Γεωργίας στην επίσκεψη στη Σλοβενία. 21 με 23 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα επίσκεψη. Πήγαμε στη Σλοβενία. Διοργανώσαμε το ταξίδι και χάρη στους συντονιστές της Επιτροπής μας και στη Γραμματεία είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τη γεωργία της χώρας μας. Η Σλοβενία, όπως ξέρετε, είναι μια μικρή χώρα. 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκτασή της. Στα χιλιόμετρα αυτά έχουμε κλίμα και υπηρετικό, έχουμε μεσογειακό κλίμα, αδριατική ακτή, που αποτελεί τμήμα της Μεσογείου και έχουμε και περιοχή των Άλπαιων. Ετοιμάσαμε το πρόγραμμα για να διαπιστωθεί η ποικιλομορφία του κλίματος. 60% της Σλοβενίας καλύπτεται από δάση. Είναι μεγάλη επιρροή των δασών στο κλίμα και 30% της έκτασης είναι αρρώσιμη γη, καλλιεργείται από το 30% το 1 τρίτο είναι αρρώσιμες γέες. 900 τετραγωνικά μέτρα αρρώσιμης γης για κάθε άνθρωπο. Άρα δεν μπορούμε να παράξουμε τρόφιμα και για άλλες χώρες και κάνουμε και εισαγωγέ κυρίως στα δημητριακά. Οργανώσαμε το ταξίδι για να δείξουμε όλα τα τμήματα της Σλοβενίας. Αυτό από τη μια, από την άλλη προσπαθήσαμε να επισκεφθούμε τους υπευθύνου για τα γεωργικά θέματα στη Σλοβενία. Πήγαμε στο Κοινοβούλιο. Ήταν καρποφόρες οι συνομιλίες με τον Υπουργό Γεωργίας. Ο Ερικάντριου ηγήθηκε της αντιπροσωπείας. Ρίκα Μίλλερ, Μάικελ Χόισλικ, ε, ο Τζέιμς Νίκολσον, η Λιδία Σέντρα Ροντρίγκε συμμετείχαν μεταξύ άλλων. Την πρώτη μέρα πήγαμε στην Eurosat Κέρσκο, Ανατολική Σλοβενία, κοντά στα σύνορα με την Κροατία, 50 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ, όπου είναι η Eurosat, ε, παραγωγή φρούτων. Μα και έχει χώρο αποθήκευσης ψυχρό, μηχανήματα διαχωρισμού καρπών και 30% των επενδύσεων ε, της εταιρεία ήταν από τους πόρους της ανάπτυξης της Πέθρου. Πήγαμε στο Χάρεκ, ανοιχτό μουσείο, παραδοσιακή αρχιτεκτονική σκίδαμε στο χωριό πώς συνδυάζουν το πρόγραμμα ε, για την ανάπτυξη Πέθρου με διάφορα άλλα προγράμματα και είναι στην κεντρική Σλοβενία η περιοχή. Φάγαμε στο Κάστρο, στη Λουμπλιάνα. Είχαμε έκθεση μελισσοκομείας. Είναι εφημισμένη η Σλοβένια για μελισσοκόμοι. 20 Μαΐου είναι η παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για τη μελισσοκομεία. Προσπαθούμε να την παγιώσουμε και γευματίσαμε με εκπροσώπους συνδικάτων, των γεωργών, εκπροσώπους συνεταιρισμών, του Υπουργείου Γεωργίας, αρμοδίου της δασοκομείας και μια ένωση γυναικών που ασχολούνται με την κελέρη της γης. Συναντήσαμε και τον Αντιπρόεδρο της Συνελεύσεως της Σλοβενίας ε, κύριο Χάιντς και τα μέλη της ε, Επιτροπής Γεωργίας, της Εθνοσυνελεύσεως, Παραγωγής Τροφίμων και Δασοκομείας και την Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνη για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πάρα πολύ καλές συζητήσεις είχαμε. Αργότερα επισκεφθήκαμε την περιοχή Πριμόρσκα που είναι κοντά στην Ιταλία και πήγαμε στην, στο αγρόκτημα Λίμπιτσα που εκεί εκτρέφονται άλογα της ράτσας Λίμπιτσα είδαμε πως ε, μεγαλώνουν τα ζώα εκεί σε αυτό το τοπίο και είναι σημαντικό και για τον τουρισμό το υποφορβείο εκεί. Και πήγαμε και στο Μπορδίβα που είναι ε, παράγει κρασί Κάβα. Πήγαμε και σε γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και κτηνοτρόφους για την παραγωγή κρέατος στην περιοχή των Άλπαιων. Παράγεται και τυρί φημισμένων και παράγεται κρέας. Όλα συνδυάζονται εκεί, τοπίο, αγροτική παραγωγή, ε, παραγωγή κρασιών. και εκεί παραγωγή ε, έχουμε παραγωγούς που είναι μέσα στους 100 καλύτερους παραγωγούς ίνων στον κόσμο στις 20 Σεπτεμβρίου το πρωί συναντήσαμε τον Υπουργό Γεωργίας, Δασοκομείας και Τροφίμων τον κύριο Ντερζίνταν και τον Υφυπουργό την Υφυπουργό κυρία Τάνια Στενίσα. Συζητήσαμε τα θέματα, την κρίση στη Γεωργία, αλλαγή του κλίματος. Είχαμε μεγάλα προβλήματα στα δάση και στην παραγωγή ίνου και φρούτων λόγω παγωνιάς, παγετού την Άνοιξη. Πήγαμε μετά στο Μπλεντ, τοποθεσία τουριστική στη Σλοβενία και έχουμε το Τρισλόσκι Εθνικό Πάρκο, το Τρίγκλο είναι το μεγαλύτερο όρος στη Σλοβενία, είναι στην περιοχή των Άλπαιων και συναντήσαμε τους αρμοδίους Το τουρμίνι στο τυρί είναι φημισμένο που παράγεται εκεί. Έχει προστασία ε, σήματος συναντήσαμε μέλη του συνεταιρισμού παρακτοτηρή και εκπροσώπους και του Εθνικού Πάρκου. Πήγαμε και στο Μουσείο Μελισσοκομείας και μιλήσαμε με των Σλοβαίνων ε, μελισσοκόμων. Ήταν και καλός και ο καιρός. Περάσαμε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τη γραμματεία και τον βοηθό μου τον Γιούρε, το ευχαριστώ επίσης, που βοήθησε να εξελιχθούν όλα ομαλά, που κάθεται μάλιστα εδώ στην τελευταία σειρά. Αν επιτρέπετε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να τοποθετηθούν μέλη που συμμετείχαν στην αποστολή, να ευχαριστήσω εν πρώτη στη γραμματεία που εξεπώνησε έκθεση, παρουσίασε την έκθεση θα πρέπει να έχετε λάβει το έγγραφο και δείχνει τον πλούτο της αποστολής, αυτών που είδαμε στην αποστολή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπόκοβιτς για την εξαντλητική παρουσίαση των όσων έγιναν στην αποστολή. Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και μέσω των συζητήσεων που είχαμε με τους διάφορους αρμόδιους θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Έρικ. Κύριε Μπόγκοβιτς, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ε, αποστολή, πολύ καλά οργανωμένο το ταξίδι, το ταξίδι συγγνώμη, εξηγήσατε τι ακριβώς κάναμε στην περιοχή και στη Σλοβενία. Στις τρεις μέρες καταλάβαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σλοβενία, αντιληφθήκαμε την κατάσταση που επικρατεί και εντυπωσιάστηκα. όταν πήγαμε στο μουσείο αυτό των ε, Σουηδών υποτών όπως το αποκαλούμε στην ε, Γερμανία μάθαμε πολλά ακούσαμε τις εξηγήσεις που μας έδωσαν οι αρμόδιοι στις διάφορες επισκέψεις που κάναμε Κύριε Μπόγκοβιτ, ήσασταν πολύ καλός που τα οργανώσατε όλα αυτά. Ευχαριστώ τα μέλη που ήρθαν μαζί μας. Γνωρίσαμε τελικά τη Σλοβενία. Ε, ήταν ένα ταξίδι στο οποίο συλλέξαμε πάμπολε πληροφορίε για τη συγκεκριμένη χώρα μέλο, Μόνο 8% της έκταξης της Σλοβενίας καλλιεργείται. Είναι αρρώσιμη γη. Ε, εξεπλάγει που τα έμαθα αυτό. και σίγουρα θα επιστρέψουμε στη Σλοβενία. Ο Αλμπερντές θα πάει με μοτοσικλέτα, είπε την επόμενη φορά. Και αν δεν υπάρχει. Αν δεν πήρατε άλογο, είναι γιατί δεν καβαλήσατε άλογο που, είχε, που δεν έγραφε πάνω BMW. Εκτός μικροφώνου, λέει ο κύριος Δέση. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι η Λουμπιάννα δεν είναι και πολύ μακριά. Είναι πιο κοντά στη, στην Αυστρία από ότι είναι οι Βρυξέλλες. Πράγματι, η κυρία Μίλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον εκ μέρου όλων των ομάδων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόγκοβιτς και σένα Έρικ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έξοχη διοργάνωση όλη την ομάδα που συνέτεινε στην επιτυχία της επίσκεψης είδαμε την ποικιλομορφία της Σλοβενίας. Τις διάφορες μονάδες που επισκεφθήκαμε, περιοχές για την προστασία της ε, ε φύσεως, ε, ε, αμπέλια, μποστάνια. Επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, πολύ ωραίο ταξίδι. Ήταν πολύ καλή αυτή η αποστολή από το πρωί, από την Ανατολή του ήλιου μέχρι τη Δύση εργαζόμασταν. Κάναμε πολλά πράγματα. Σε δυόμιση μέρες είναι απίστευτο το πόσα πράγματα κάναμε. Ήταν έξοχες οι συζητήσεις με τους πολιτικούς, με τους υπουργούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσβλέπω σε μια άλλη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσω μόνη μου στη Σλοβενία. Ευχαριστώ ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρέπει να πούμε ότι είδαμε το αντίστοιχο της BMW του Albert στη Σλοβενία. Ε, το ξέρουμε και πόσο γρήγορα ταξιδεύει στους αυτοκινητόδρομους γερμανικούς. Ευχαριστούμε όλους για τη διοργάνωση. Και ο Μπέγκοβιτς ήταν πολύ καλή φιλοξενία σας. Ε, ήταν άκρος εκπαιδευτική επίσκεψη. Η Σλοβενία προχώρησε πολύ. Έχει ακόμα δρόμο να κάνει, πιθανότατα, αλλά εύχομαι σε όλους καλή τύχη και ευημερία στο μέλλον. Πολλές ε, ευχάριστες αναμνήσεις έχω από τότε. Αποδεικνύεται η ανάγκη που έχουμε εμείς τα μέλη της Επιτροπής να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε επί τόπου τι γίνεται. Να, να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές, πέρα από αυτές που γνωρίζουμε εμείς τις δικές μας. Ε, έτσι θα είμαστε και καλύτερα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα διάφορα προβλήματα. Είναι πολύ ποικιλόμορφη η Ευρώπη από βορρά στο νότο, ανατολικά, δυτικά, μεγάλες διακυμάνσεις τοπίων και κλίματος. Και κυρίως είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι. Θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια επιστροφή σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίκολσα. Ο κύριος Άγνη τώρα. Yes, Κύριε Άγνιου, εγώ δεν πήγα στη Σλοβενία, αλλά πήγα στο Κόρκ, στην Ιρλανδία, για μια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί συνάντησα ένα νέο Σλοβαίνο αγρότη και μου είπε κάτι που με ευνηδίασε. Μου είπε ότι πολλοί νέοι αγρότες ε, φεύγουν από τη Σλοβενία ή αν δεν φεύγουν από την Σλοβενία τουλάχιστον αγοράζουν αγροκτήματα στη Σερβία που δεν είναι καν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν πρόσβαση στη ρωσική αγορά. Το επιβεβαιώνει ή το διαψεύδει αυτό ο κύριος Μπόγκοβιτς. Επίσης, ε, τι γίνεται με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις στη Σλοβενία. Έχουμε παγωνιές, παγετούς, ε, αργά προς, την, προς το τέλος της Άνοιξης και φαίνεται ότι παρατράβηξαν οι προσπάθειε μα να αναχαιτήσουμε την αναθέρμανση του πλανήτη αρκετά πια. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Η κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδος μου τον Έρικ για την ε, πολύ καλή οργάνωση αυτής της αποστολής. Και αν ποτέ χάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να γίνεις τουριστικός οδηγός, ξεναγός γιατί είσαι εξαιρετικός στην ξενάγηση. Απίλαψα πραγματικά αυτό το ταξίδι στη Σλοβενία. Γιατί ναι μεν ήταν ταξίδι για εργασία, αλλά εγώ παρόλα αυτά διασκέδασα και όλο το απόλαυσα και εξοικειώθηκα κάπως με την Σλοβενία, το καταπληκτικό αυτό κάστρο ήταν στο επίκεντρο αυτής της ε, αποστολής. Εργαστήκαμε ε, ακαταπώνητα, αλλά διασκεδάσαμε και όλα περάσαμε πολύ καλά και χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι ε, κάνεις μεγάλη προσπάθεια στην περιφέρειά σου, είσαι πασίγνωστος εκεί, είχαμε επαφές με πολύ κόσμο και μάλιστα εντυπωσιάστηκα από τον ε, Υπουργό Γεωργίας της Σλοβενίας που μιλούσε γερμανικά άπτεστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή, κατατοπιστική και πολύ ενδιαφέρουσα η επαφή που είχαμε με πολιτικούς ηθήνοντες ε, για τη Γεωργία Υψηλή επίπεδου. Σίγουρα δεν ήταν ταξίδι αναψυχής, παρόλο που ήταν πολύ ευχάριστο. Αλλά ήταν ε, ταξίδι εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι να πω, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μπόγκοβιτς για τη φιλοξενία που μας πρόσφερε για την άρτια οργάνωση της αποστολής και για όλες τις συζητήσεις ε, που είχαμε. Έτσι, εξοικειωθήκαμε κάπως με την ε, Σλοβενική Γεωργία, κυρίως της Ανατολικής ε, Σλοβενίας και ανταλλάξαμε απόψεις για θέματα που μας απασχολούν όλους, το θέμα της υγιής, των γεωργικών τιμών, τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα. Πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποστολή και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή την άγουσα να ακολουθούμε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν Χόισλινγκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Μπόγκοβιτς γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή αυτή και πραγματική απόλαυση αυτή η επαφή με την ε, Σλοβενία και τις περιφέρειές της. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πόσος κόσμος ζει από τη γεωργία. Με μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μέσο όρο 8 εκτάρια αναγεωργική εκμετάλλευση. Και είδαμε τις προσπάθειες ε, των γεωργών να διαφοροποιήσουν κάπως ε, το γεωργικό του εισόδημα προσθέτοντας και τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό στις δραστηριότητές τους και σίγουρα τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα έχουν επενδυθεί θαυμάσια στη Σλοβενία που είδαμε πόσο καλά αξιοποιούνται και πόσο δημιουργούν προοπτικές για το μέλλον. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ φιλοευρωπαϊκό το κλίμα στη Σλοβενία και οι Σλοβαίνοι πολίτες στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά τουλάχιστον είναι φιλοευρωπαίοι. Ευχαριστώ. Ο Φραντς Μπόγκοβιτς και πάλι. Σας ευχαριστώ. Πολύ ευγενικά τα λόγια σας. Ε, να απαντήσω στον κύριο Άγνιο. Καταρχήν ελπίζω ότι στην επόμενη ε, συνάντηση, στην επόμενη αποστολή θα μας συνοδεύσετε. Στην Σλοβενία έχουμε περίπου 70.000 ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ενεργούς γεωργούς, με ανθρώπους δηλαδή που βιοπορίζονται από τη γεωργία, που εξαρτώνται για το βιοπορισμό τους από τη γεωργική παραγωγή. Στη χρηματοοικονομική περίοδο 2007-2010 είχαμε περίπου 4.000 νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για τους νέους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό τμήμα της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, ιδιαίτερα του σκέλους ανάπτυξης πέθρου. Και μάλιστα, όπως είπε ο κ. Μάρτιν, έχουμε μικροκαλλιέργειες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με διαφοροποίηση. Και αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρής ε, κλίμακος είναι η απάντηση ίσως στα προβλήματα που έχουμε με τη γεωργία. Και χρειαζόμαστε φυσικά αυτό το νέο αίμα στην Σλοβενική γεωργία. Ο συνολικός αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να μειώνεται, αλλά ακριβώς εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής μας στην κοινή γεωργική πολιτική, έχουμε κάπως αναχαιτήσει αυτή τη μείωση ε, του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχουμε όλο και περισσότερες και πιο άμεσε επαφές μεταξύ παραγωγών, καλλιεργητών δηλαδή και καταναλωτών, κάτι που ε, επιτρέπει την επιβίωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τώρα για την αγορά ε, κτημάτων από Σλοβαίνου στη Σερβία, αν παρακολουθήσουμε τις εξαγωγές ε, από την Σερβία προς τη Ρωσία, από την Λευκορωσία και το Καζακστάν προς τη Ρωσία, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι διέξοδοι στο μέτρο που ισχύει το εμπάργο το ρωσικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν το αρνούμε, αλλά το βασικό είναι να παραμείνουν οι νέοι στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. και εγώ είμαι μιλοπαραγωγό και εγώ υπέφερα φέτος, γιατί είχαμε παγετός 26 Απριλίου, αργά την Άνοιξη, και πολλοί καλλιεργητές ε, οποροφόρων δέντρων είχαν πρόβλημα και ενώ η μέση παραγωγή ήταν 120 με 130 τόνοι το χρόνο, φέτος είχαμε μόνο 14 τόνους εξαιτία του όψιμου παγετού. Και είχαμε πολλούς οπορώνες ε, με προστασία με τα δίκτυα. Είχα και εγώ ε, αρδευτικά συστήματα στους απορώνες μου με τη στάγδιν άρδευση, με πολύ μικρή χρήση νερού για την άρδευση. Και ε, όπως το είπε και χθες η Μαριάννα Πετήρ και η Κροατία προβληματίστηκε και ε, επλήγει από αυτό το θέμα της ε, έλλειψης του νερού και τα συστήματα προστασίας κατά του παγετού είναι τόσο ακριβά, τόσο δαπανηρά που ο κόσμος προτιμά να μην τα χρησιμοποιήσει. Και όμως σώζουν κάτι τέτοια συστήματα. Χάνονται δυστυχώς ε, πολύτιμοι πόροι νερού. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για τα συστήματα προστασίας από τον παγετό. Πάντως αυτό που προσπάθησα να δείξω με αυτό το ταξίδι για την αποστολή στη Σλοβενία είναι να σας δώσω να καταλάβετε ότι απαιτείται η σύνδεση της ζωής της πόλης ε, και η να τη συνδυαστεί με τη ζωή στην Ήπεθρο. Για να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια για την ανάπτυξη Ήπεθρου με άλλα περιφερειακά κονδύλια και κονδύλια συνοχής. Γιατί, όπως είδατε, το βιωτικό επίπεδο στην Ήπεθρο σε πολλά τμήματα της Σλοβενίας είναι παρεφερές με αυτό των πόλεων γιατί μπορεί να υπάρχουν και εκεί προβλήματα ανεργία στην Ήπεθρο, αλλά δεν είναι πολύ χειρότερο το βιωτικό επίπεδο από ό,τι στι πόλει. Το βασικό είναι οι νέοι να παραμείνουν στην Ήπεθρο και υπάρχει η δυνατότητα μετακίνηση. Και στις, στο πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 συνδυάσαμε πολύ καλά τα διάφορα είδη κοινοτικών κονδυλίων και το εκτιμά ιδιαίτερα και ο λαός γιατί είδε αποτελέσματα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Γι' αυτό και η κοινή γνώμη είναι πιο θετική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αγαπώ τη χώρα μου και το σχόλιο σα να γίνω ξεναγός αν μείνω χωρίς δουλειά <laughs> το εκτίμησα ιδιαίτερος γιατί πραγματικά αγαπώ την πατρίδα μου. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Όντως, ήσουν ε, εξαιρετικός ξεναγός στην αποστολή. Νομίζω ότι είδαμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που είπες για την διαφοροποίηση της γεωργίας, ε, που την είδαμε με τα μάτια μας στη Σλοβενία. Και επίσης είδαμε πόσο σημαντική ήταν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδαμε και επιτόπου την πρόσφατη ιστορία της Σλοβενίας και μετά την ανεξαρτοποίηση. Είδαμε σε πόσο λίγο χρόνο κατάφερε ο κόσμος να προσαρμοστεί, ε, να δείξει τέτοιο επαγγελματισμό, να ε, δείξει αλληλεγγύη και να προχωρήσει τόσο πολύ. Είδαμε πόσο ε, σημαντική ήταν η δυναμική της Σλοβενίας στη Γεωργία και είναι υπόδειγμα η πρόοδος που συντελέσατε στη χώρα σας στα θέματα αυτά και ευχαριστούμε και τη Γραμματεία για την πολύ καλή οργάνωση. Ήταν πραγματικά άρτια αποστολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Προτείνω τώρα να συνεχίσουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση για την απαλλαγή του 2015. Ο Άλμπερ pardon. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε το 11 πρώτα και το 10 μετά. Διότι ο κύριος Γιάρη είναι ακόμα στην άλλη επιτροπή. Διαφορετικά θα ασχοληθώ ίσως εγώ με το θέμα. Κατά τον ενημερώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε το πρόβλημα ότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προπολογισμό. Θα μπορούσες, ενδεχομένως θα μπορούσατε, λοιπόν εσείς κύριε Ντάς, να τοποθετηθείτε στη θέση του κυρίου Ζάρ, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Θα προτιμούσα να κάνουμε αυτό για να εκμεταλλευτούμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε θα μπορούσε να τοποθετηθεί για την απαλλαγή του 2015. Αν συμφωνείτε, θα προτιμούσα αυτό να κάνουμε. Καλώς, ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Ντες, ο Πίτερ Γιάρ μου έδωσε την άποψή του, θα παρουσιάσω τι λέει, υποβολή τροπολογιών, η προθεσμία είναι 5 Δεκεμβρίου. Ψηφοφορία πιθανότατα στην Επιτροπή 25 και 26 Ιανουαρίου του χρόνου. Βασικά σημεία των ε, γνωμοδοτήσεων για το 2015 είδαμε 2,9% μείωση αύξηση, αύξηση σε σχέση με τον περσινό χρόνο. Μάλλον το ποσοστό σφάλμα, ποσοστό σφάλματος 2,2% στον πρώτο πυλώνα, χαμηλό ποσοστό σφάλματος, πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε στο δεύτερο πυλώνα, 5,3%. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε περισσότερο αυτά που συμβαίνουν στο δεύτερο πυλώνα, τα σφάλματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν είναι σφάλματα όσον αφορά τα δεδομένα για τη χρήση των διαφόρων επιφανειών. Δεν μιλάμε για απάτες, δεν είναι πρόβλημα απάτης, δεν είναι πρόβλημα σπατάλης δημοσίων χρημάτων, απλώς λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων που αφορούν τις ε, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχουμε διάφορα είδη σφαλμάτων, άμεσες πληρωμές, Φερρυπίν. Είναι τέσσερα είδη σφαλμάτων εκεί. Ένα, χωρίς μια κατηγορία χωρίς αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Μετά, διαφθορά, μεγάλη διαφθορά. Αυτές είναι οι κατηγορίες που πρέπει να υποδιαρέσουμε τα σφάλματα εν γέννη. Κάποια σφάλματα δύο τετραγωνικά εδώ παραπάνω, δύο λιγότερα δεν θα καταστραφούμε. Ο κύριος Γιάρ καλωσόρισε τις διάφορες δραστηριότητε της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας που εξέτασε τα θέματα της κοινή αγροτικής πολιτικής και τους διάφορους τομείς παραγωγής τροφίμων. Καλωσορίζει επίσης ότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται ανάλυση των σφαλμάτων με νέα προσέγγιση. Και πάμε και στον ίδιο, ο οποίος κατέφτασα. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Είχα ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναφορών, βλέπετε, και είμαι συντονιστή εκεί. Και δεν μπορούσα να φύγω. Τα καλά μαντάτα α... υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλα καλά μαντάτα. Υπάρχουν και κάποια άσχημα. Στους Κιώδης έγινε μια πρώτη συζήτηση. Την περασμένη Τετάρτη στο Στασβούργο έγινε η συνεδρία των Σκιωδών. Το είχα προτείνει αυτό, αλλά η διοίκηση δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ έστειλα διαμαρτυρία στον πρόεδρο για αυτό το λόγο. Δεν είναι καλό αυτό που έγινε. Καμιά φορά σε χρόνους ειρήνης η δίκηση αντικαθεστά τον εχθρό. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ η δίκηση. Η δίκηση λοιπόν του Κοινοβουλίου, δεν μιλάω για τη γραμματεία, μιλάω για τη δίκηση του Κοινοβουλίου, δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει τις εργασίες, όπως δεν μας επέτρεψε να κάνουμε τη συνεδρίαση των ε, σκιωδών και ακύρωσε τη συνεδρίαση των σκιωδών, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πράγματα να συμβαίνουν Ίσως να είναι πολύ παραδοσιακό εδώ, αλλά είναι κάτι ανέφικτο σε εθνικό επίπεδο. Ήταν καλή ημερομηνία αυτή. Ε, είχαμε όλου του κοιόδη στο Στρασβούργο, είχαμε την αίθουσα, είχαμε του διερμηνεί και τελικά ακυρώθηκαν όλα. Λόγω δίκηση. Δεν δόθηκε συνέχεια τελικά. Υπάρχουν και αναβολέ. Αυτό είναι λυπηρό. Θα διαμαρτυρηθώ περαιτέρω και λέω ονόματι όλων ότι δεν είναι κάτι που μας βόλεψε θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το θέμα να δούμε ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά. Αλλά είναι σημαντικό να γίνεται συνεδρία στους σκιωδών, γιατί βελτιώνεται και η ψηφοφορία και η έκθεση. Αυτά ήταν τα κακά μαντάτα. Λοιπόν, τελικά συνέβη αυτό, το θεώρησα απίστευτο αυτό που μας ακύρωσαν τη συνεδρίαση. Ίσως ο, ο πρόεδρος θα λάβει πληροφορίες, θα πρέπει να μάθουμε. Αν θεωρούν οι βουλευτές ότι χρειάζεται συνεδρίαση των σκιωδών, θα πρέπει τελικά να λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεδρίαση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντές, ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ξεκινάμε λοιπόν. ο κύριος Μπέλντερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιάρ, έξοχη γνωμοδότησή του, όσον αφορά την απαλλαγή. Κάποια σχόλια να επιτρέπετε συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε. Η παρουσίαση που αφορά τον πρώτο πυλώνα. Είπατε ότι το σφάλμα είναι 2,2% το ποσοστό σφαλμάτων στον πρώτο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα το ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο από ότι στον πρώτο πυλώνα. Άρα είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, επιδόσεις στους διαφορετικούς πυλώνες. Καλό θα ήταν αν το ελεκτικό συνέδριο στο μέλλον συνεχίζει να μας δίνει στοιχεία και τους δύο πυλώνες ξεχωριστά. Το ποσοστό σφαλμάτων για τους δύο πυλώνες. Είναι καλό που θα συνεχίσουν, αν συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον αυτό. Μετά ανάπτυξη υπαίθρου. Απλουστευμένες επιλογές όσον αφορά το κόστος. Ε, αυτό ίσως οδηγήσει σε λιγότερα σφάλματα. Απλουστευμένη κοστολόγηση ίσως οδηγήσει σε χαμηλότερα σφάλματα. Και συνεισφορές κατά αποκοπήν ή τιμές μονάδας τυπικές. Οι συνεισφορές κατά αποκοπήν ή ε, τυπικές ε, τιμές μονάδας. Ε, αυτό θα απλούστευε τα πράγματα και θα ενδυνάμωνε την επιχειρηματικότητα. Τέλος, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο εξακολουθούν να εξετάζουν τους δείκτες επιδόσεων με βάση το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο εξετάζουν τον προπολογισμό βάση επιδόσεων. Αυτό είναι σωστό για την καινοτομία. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την άποψή του, για την γνωμοδότησή του. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί ε, στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπέλντερ. Η κυρία Σένερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση μόνο και δεν ξέρω αν μπορεί να μου εξηγήσει ο εισηγητής σε ποια προγράμματα ε, μικρότερων οδοτήτων ε, εννοεί και προτείνει την μετάβασή του στον δεύτερο πυλώνα. Για το σημείο 6 θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Ο κύριος Βιέγκας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω κάτι διαφορετικό. Και δηλαδή, δείτε, σε σχέση με αυτά τα οποία ελέγχθησαν για την ε, συνάντηση των ε, σκιωδών συγητών το Στρασβούργο. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσαμε ενδεχομένω να γίνονται κατ' εξαίρεση την εβδομάδα της συνεδρίασης ε, συνεδριάσης αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε πολύ πιο σημαντικά θέματα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίες. Νομίζω ότι κάθε τέσσερις εβδομάδες πάμε σε ολομέλεια και βεβαίως αυτό το οποίο θα πρέπει κυρίως να τονίζουμε και δίνουμε προτεραιότητα είναι στη συνεδριά της ε, Ολομελίας. Έχουμε τρεις εβδομάδες μεταξύ των ολομελιών για να ασχοληθούμε με τις άλλες συνεδριάσεις και με τα άλλα μας θέματα. Δεν θα πρέπει να παραφορτώνουμε μια ήδη πάρα πολύ φορτωμένη μερίστια διάταξη της ολομελίας. Βεβαίως, υπάρχουν και εξαιρετικές έκτακτες καταστάσεις Απλώς θα ήθελα να τονίσω αυτό. Η δική μας αρχή πρέπει να είναι ότι στα πλαίσια του δυνατού δεν θα πρέπει να αναλωνόμαθε σε συνεδριάσεις και οδών εισηγητών, συνεδριάσεις επιτροπών. Θα πρέπει κυρίως να ασχολούμεθα με την Ολομέλεια δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα για τα οποία πρέπει να αποφαίνομαστε. Τώρα σε σχέση με την έκθεση αυτή επί τη ουσία θα ήθελα να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία λέγεται, κυρίως σε σχέση με το ποσοστό φάσμα, το στο οποίο είναι αρκετά διαφορετικό στον πρώτο ή δεύτερο πυλώνα και να πω ότι θα πρέπει εμείς να υπογραμμίσουμε ότι είναι πάντα αναγκαίο να υπεραπλουστεύουμε διότι Πολλές φορές βλέπουμε ότι κυρίως σε θέματα δαπανών δεν έχουμε πάντα το σωστό ποτό στη σωστή θέση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το ποσοστό σφάλματος ίσως. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις δημόσιες συμβάσεις, τις προμήθειες, όπως μας επισημαίνει και το λυτικό. Ναι, τώρα, νομίζω όλο και περισσότερο τα δημοσιονομικά ε, είναι κάτι το οποίο, μέτρα είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βλέπουμε στην ΚΑΠ. Αλλά το θέμα αυτό θέτει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την ε, συνοδευτικά μέτρα και τον έλεγχο τον οποίο πρέπει να κάνουμε, δεδομένου ότι εγείρονται διάφορα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σχέση με το θέμα αυτό. Τώρα, για να ολοκληρώσω. Βεβαίως αυτό που μας απασχολεί κυρίως δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο απολογιστικής πλευράς θα δούμε πώς ε, αναπτύσσονται οι λογαριασμοί. Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται τα κονδύλια της ΚΑΠ ώστε να μπορέσουν κάποιες καλλιέργειες να επωφεληθούν και να δούμε πώς θα αποφύγουμε την μη δίκαιη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων, κυρίως για να μην επιβάλλουμε κυρώσεις στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτά είναι μια κριτική την οποία θα ήθελα να κάνω και κυρίως επί της ουσίας να πω ότι τα ευρωπαϊκή θεσμή, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να δουν πώς θα κάνουν ε, περαιτέρω φιλελευθερωποίηση της ΚΑΠ και όπως ξέρετε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση και με τον κοινοτικό προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε αυτή την κατανομή που κάνουμε πάντα πολύ πιο προσεκτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόταση αυτή που είναι καλή στην έκθεση που μας παρουσιάσετε. Αρχίζοντας θα ήθελα να πάω το 2015, ήταν πρώτο έτος πλήρους <laughs> εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, κυρίως όσον αφορά τις συμφωνίες επιπλωμών. Επίσης, είναι τότε και η έγκριση των νέων προγραμμάτων ανάπτυξης για τη νέα περίοδο. Είναι καλές οι προτάσεις που γίνονται με τη γενικότερη πρόταση συμφωνώ. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εξεργαστούμε περαιτέρω. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και κάποια σημεία πολύ σημαντικά που θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το γεγονός ότι το ποσοστό ε, σφάλματος ε, έχει φτάσει σε 2,2 ενώ στο παρελθόν είχαμε ποσοστό 3,6. Επίσης, ζητείτε ε, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για να μπορούμε να ελέγχουμε τις απάτες για να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος δεδομένου ότι και πάλι έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος γύρω στο 2%. Έχω για το σημείο 6 κάποιες πληροφορίες να ζητήσω όπως και άλλοι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται με μεγάλη ακρίβεια ώστε ή να καταθέσουμε τροπολογίες ή να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην πρόταση. Τώρα, όσον αφορά την περαιτέρω αξιολόγηση των κοινωνικών ε, οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ήπεθρος είναι κάτι πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια κοινή αξιολόγηση και να έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινούμεθα και καταδεικνύουμε δείκτες για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση με από κοινού ε, ε, μελέτη και από τα κρατημέλη και από την Κομισιόν. Θα πρέπει να είμαστε όμως υπερήφανοι και να πούμε ότι μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτής της πολιτικής να παρέχει και μία ε, πολιτική ε, τροφίμων η οποία να είναι υψηλού επίπεδου. Η απλοποίηση είναι κάτι που βοηθάει. Θα θέλαμε και περαιτέρω απλοποίησης. Και είδαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ε, έγγραφα πρέπει να συμπληρώσει κανείς, έγινε μια επίδειξη γι' αυτό, για να μπορέσει να έχει κάποια κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν η προσέγγιση μας να είναι πάρα πολύ πραγματιστική όσον αφορά τις, τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται και δαπανώνται τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για την ΚΑΠ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα υποστηρίξουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάρεν Κάλεμπαχ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντες που κατέθεσε την έκθεση αυτή και τον κύριο Γιάρ που την παρουσίασε. Πιστεύω ότι οι συναντήσεις συνταξή και οι η εισηγητών είναι πολύ σημαντικές, ίσως όμως δεν είναι ιδανικός τόπο το Στρασβούργο για τέτοιου συνεδριάσεις, γιατί έχουμε και πολλές άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πολύ συχνά οι συνεργάτε μας, οι οποίοι χειρίζονται τους φακέλους αυτούς, δεν είναι και πάντα διαθέσιμοι. Θα πρέπει να είναι λοιπόν μια εναλλακτική λύση ίστατη το Στρασβούργο. Όταν έχουμε να χειριστούμε ένα θέμα κατεπήγων. Διαφορετικά θα πρέπει εδώ στις Βρυξέλλες να οργανώνονται συνείδριασεις. Βλέπουμε ότι το ποσοστό σφάλματος μειώνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο το οποίο θα αναφέρω. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα υψηλό ποσοστό σφάλματος δεν σημαίνει πάντα απαραίτητος ότι δεν χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια του Ευρωπαίου φορολογούμενου ή ότι υπάρχει διαφθορά απαραίτητο. Πολλές φορές αυτό μπορεί να καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην δίκηση. υπάρχει επαχθής γραφειοκρατία, υπάρχουν άλλου είδους εμπόδια και προβλήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί επίσης και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και τα τελευταία χρόνια και στα κράτη-μέλη και από το ελεγκτικό συνέδριο και νομίζω ότι τώρα και τα κράτη-μέλη έμαθαν να κάνουν ε, εξέταση όλων των μεγεθών στα οποία θα μπορούσε να υπησέρχεται σφάλμα. Έχουν βελτιωθεί οι μέθοδοι και το ότι ε, ε, περάσαμε σε ποσοστό σφάλματος από 3,6 στο 2,9 είναι θετικό. Αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς διαμορφώνεται η γενική κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με το μικρότερο ποσοστό σφάλματος στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Και τα κράτη-μέλη την πράξη είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των ε, δαπανών, αλλά θα πρέπει να προσθέσω και το εξής. Το Ελεκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφεραν διαφορετικά ποσοστά σφάλματος. 5,3 για την ανάπτυξη της Ισπέθρου. Ίσως διότι ακολουθείται διαφορετική μέθοδος. Θα πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε σε εναρμόνιση ενδεχομένως και αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι δουλεύουν σωστά όλα τα πρότυπα ε, ελέγχου που γίνεται με σφιγμομέτρηση 180 έλεγχοι έγιναν εκ μέρους της Επιτροπής και αν το δείγμα που χρησιμοποιούμε είναι σωστά επιλεγμένο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν θα πρέπει όμως ε, να επιτρέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό σφάλματος για να μην έχουμε περισσότερες ε, δαπάνες αν πρέπει συνέχεια να κάνουμε ελέγχους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να προσπαθούμε να δουλεύουμε με διαφορετικούς δείκτες δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων τα οποία κάποια στιγμή δεν χρησιμεύουν σε τίποτα Κάποιες φορές έχουμε δείκτη για να μετρήσουμε πόσα ε, είναι ποιο είναι το ύψος της κάθε μιλιάς, πόσα μήλα μας δίνει κάθε μιλιά. Στην ε, κτηνοτροφία μιλάμε για διάφορα δείκτες που αφορούν την πυκνότητα των ε, ζώων ανα περιφέρεια, περιοχή. Έχουμε κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με πιο ενίο τρόπο. Όσον αφορά τα καταποκοπήν ποσά, θα πρέπει να τα εξετάσουμε διότι διαφορετικά θα μπούμε σε λεπτομέρειες λογαριασμών και θα ψάχνουμε τα μικρά ευρώ ή τα, το 50 λεπτά του ευρώ για να δούμε πώς θα κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των μεγεθών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πολλές φορές γίνονται υπολογισμοί οι οποίοι δεν είναι και τόσο χρήσιμοι. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφέρω. Είναι λογικό το ποσοστό σφάλματος, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε πολύπλοκα προγράμματα μειώθηκε, μάλλον μειώνεται ε, κάθε χρόνο και περισσότερο το ποσοστό σφάλματος παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε να κάνουμε με απολύτως αξιόπιστο στοιχείο εδώ. Στο σημείο 4 λέει ο συνάδελφος ότι δεν υποβάλλονται ε, σωστά οι εκθέσεις από τα διάφορα κράτη. Έχουν όμως τη δυνατότητα αν καλυφθεί ότι υπάρχουν σφάλματα να αλλάξουν τα στοιχεία. Θα ήξερα το σημείο έξι να το διαγράψουμε διότι πιστεύω ότι τα πολύ μικρά προγράμματα του πρώτου πυλώνα δεν θα πρέπει να μεταφερθούν, μεταφερθούν στον δεύτερο, διότι εδώ τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης και θα αυξηθεί το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Έχω και κάποιες άλλες προτάσεις για τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσω αργότερα και θα ήθελα να ζητήσω και το εξής. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και έχω Στην σελίδα 8 στο σημείο 15 κάποιο πρόβλημα. Γίνεται λόγος για κάποια ε, προβλήματα στο PIS, κάποια σφάλματα και μιλούμε για landfill. Αλλά δεν είναι landfill, land parcels. Δεν μιλούμε δηλαδή για κάτι το οποίο αφορά τα, ε, την αποκομιδή των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα είχα ερωτήσεις να θέσω, πολύ απλοϊκές, αλλά αναφέρθηκε ο συνάδελφος προηγουμένως αυτό. Πρέπει να πω ότι για τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός είναι άγνωστο έδαφος ακόμα για μένα. Έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό το ποσοστό σφάλματος τι είναι. Θα ήθελα έναν ορισμό του ποσοστού σφάλματος. Θα μπορούσατε ίσως να μου στείλετε κάτι στο γραφείο μου. Ε, οι άλλοι σου ξέρουν, εγώ δεν γνωρίζω, θα με ενδιαφέρε να μάθω. Τι γίνεται με το ποσοστό σφάλματος, αναπρόγραμμα. Υπάρχει διαφορά επίπεδου σφάλματων στο δεύτερο πυλώνα από ότι στο πρώτο. Το ποσοστό σφάλματος σχετίζεται με ένα οικονομικό ποσό συγκεκριμένο. Πρόκειται περί ενός ποσοστού, το καταλαβαίνω βέβαια αυτό. Δύο χρόνια είμαι στο Κοινοβούλιο και ακόμα χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος, ποιος είναι ο ορισμός του ποσοστού σφάλματος. Διότι εδώ μοιάζει σαν να προσπαθούμε να συγκρίνουμε μήλα με χλάδια. Ο κ. Νταντέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα, αρκετά πρόσφατα, συνομίλησα με τον νέο Πρόεδρο του ελεκτικού Συνεδρίου. Πρώην συνάδελφος, είναι, που ήταν πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία. Ένα ελεκτικό συνέδριο κάνει προσταφαιρέσεις και ελέγχει. Στη Γεωργία όλος ιδιαίτερος χρειαζόμαστε ποιοτική εξέλιξη των εκθέσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο έχει χιλιάδες υπαλλήλους τους έχει αποτελματώσει λόγω ατελών χαρτοφυλακίων χωρίς να εξετάζει κατά πόσο ο στόχος των προσπαθειών ήταν σωστός ή όχι. Οι δαπάνες έγιναν. Οι δαπάνες που έγιναν παρήγαγαν αποτελέσματα που ακολουθούν την πολιτική που ελέγχεται ή όχι. Αυτό το ξέρουμε. Αυτή η πολιτική του ελεκτικού συνεδρίου, η έλεγχη που διενεργεί το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να μας οδηγούν σταδιακά στο να μπορούμε να κρίνουμε ε, το πόσο βάσιμες είναι οι πολιτικές μας, πόσο χρήσιμες. Και όχι να βλέπουμε αν ένα θέμα έχει ολοκληρωθεί, είναι πλήρες ή όχι, ένα χαρτοφυλάκιο είναι πλήρες ή όχι. Θα πρέπει το ελεκτικό συνέδριο να εξετάσει και ποια είναι η σύνθεση των διαφόρων προγραμμάτων και των χαρτοφυλακίων. έχουν ε, προσθέσει διάφορες, στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης διάφορες στιβάδες στην πολιτική. Στην προηγούμενη μεταρρύθμιση είδα όταν εφαρμόστηκε, όταν πηγαίνω επί τοπίου, ε, τελικά όταν έχουμε εφαρμόσει διάφορα προγράμματα πηγαίνει επί τόπου, τελικά έχει αλλάξει η μορφή. Ο καθένας έχει προσθέσει για να προστατευτεί κάποια, ε, κάποια στιβάδα παραπάνω. Θα πρέπει αυτή την παραποίηση της παραγωγής που θέλαμε να την καταπολεμήσουμε. Διότι η νομιμότητα μιας πολιτικής είναι αυτή που θεσπίζουμε εμεί και όχι τις πολιτικές που εφαρμόζεται αφού ο καθένα προσπαθεί να προστατευτεί. Θα πρέπει να μα βοηθήσει ε, το ελεκτικό συνέδριο στη δουλειά να ελέγχουμε τα αριθμητικά στοιχεία να πηγαίνουν πιο πέρα από τον απλό έλεγχο των αριθμητικών στοιχείων. Στην τελευταία μεταρρύθμιση συλλογικά θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μαζί με εμά, όταν σε μια χώρα οι έλεγχοι που διενεργούνται δείχνουν ότι το, μειώθηκε το ποσοστό να μπορούμε να μειώνουμε τους ελέγχους που γίνονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Την επόμενη έκθεση θα ήθελα το ελεκτικό συνέδριο να μας δείξει πώς εφαρμόζεται αυτή η ελάφρυνση των ελέγχων. Διότι είμαστε στο τέταρτο έτος της γεωργικής πολιτικής υπό τη νέα μορφή που έχουμε θεσπίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι διαιρείται σε δύο αυτή η συζήτηση. Υπάρχει ένα θέμα καταρχήν τακτοποίηση ε, και ε, τα του, των, των πραγμάτων του οίκου μας, ε, τα διαχειριστικά και το δημοσιονομικά. Ε, την Δευτέρα το απόγευμα συνήθως μιλάω στην Ολομέλεια, γι' αυτό, από αυτό εξαρτάται έθιμη περί κατά μιας έκτακτης συνεδρίασης. Πώς ε, θα αντιδρούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν λέγαμε ότι θα είχαμε συνεδριάσεις ε, την Παρασκευή το απόγευμα μετά την ψηφοφορία. Δεν νομίζω να περνούσε εύκολα μια τέτοια πρόταση. Και υπάρχει και ένα εγχειρίδιο κανόνων που προβλέπει ότι το Στρασβούργο και ελπίζω να με προσέξει ο Φιλίπ, γιατί φαίνεται ότι κυρία αλλού. Γνωρίζει τον ε, κανονισμό ο Φιλίπ, που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται διοργάνωση συνεδριάσεων επιτροπών στο Στρασβούργο. Α το λάβουμε υπόψη και επίσης λέμε που, που κατασπαταλούνται κονδύλια και που χάνονται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουμε τεράστιες προσπάθειες ακριβώ ε, ακριβώς για να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια και να μην πηγαίνουν χαμένα. Κάνουμε τέτοια προσπάθεια ε, και είναι τόσο χρονοβόρα διαδικασία που τελικά μας ε, βάζει πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστερημένη καταβολή των πληρωμών. Και να ένας επιπλέον πολύ καλός λόγος υπέρ του Brexit. Ευχαριστούμε κύριε Άγγινιο. Ο κύριος Φλάναγκαν. Μιλάτε για το υψηλό ποσοστό σφάλματος του δεύτερου πυλώνα. Είχαμε μια έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού της 20... του 2014 που εστιάστηκε στο δεύτερο πυλώνα και ένα από τα προβλήματα ήταν ο κανονιστικός υπερθεματισμός, το gold plating σε εθνικό επίπεδο. Ένα από τα προβλήματα του δεύτερου πυλώνα ήταν η περιπλοκότητά του. Ήταν ανέκαθεν πιο περίπλοκο ο δεύτερο πυλώνα. Τώρα προσπαθούμε να πλουστεύσουμε κατά προτεραιότητα τον πρώτο πυλώνα. Ενώ είναι προφανέστατο ότι το βασικό πρόβλημα πολυπλοκότητα το φέρει ο δεύτερο πυλώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα οργανωτικά. Την τελευταία φορά ε, είχαμε σύμπτωση των συνεδριάσεων τη δική μα επιτροπή με τι επιτροπέ Ελέγχου Προπολογισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και προσπαθούσα να τρέξω από τη μία ε, συνεδρία στην άλλη για να προλάβω τι παρουσιάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη μία και στην άλλη επιτροπή. Όταν έφτασα στην συνεδρίαση, ο αρμόδιος ηγητής της απαλλαγής έλεγε τι κρίμα που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες οι ενδιαφερόμενοι. Μα δεν μπορούμε να είμαστε παντάχου παρόντες, να είμαστε παρόντες ταυτόχρονα σε δύο συνεδριάσεις όταν συμπίπτουν. Και σε ό,τι αφορά το επιχείρημα ότι είναι ο γεωργικό προπολογισμό ο, ο μεγαλύτερο και δεν γίνεται σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων, θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη διοργάνωση ώστε να μπορούν να πηγαίνουν οι συνάδελφοι και στι ε, δύο συνεδριάσει και των δύο επιτροπών. Επίση, ο κύριο Ζέλλερ είπε ότι ε, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του και είναι μέρος του ΕΛ και αυτό με προβληματίζει είναι ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους ε, μεγαλοκαλλιεργητές και μάλιστα η βασίλισσα της Αγγλίας είναι από τους μεγαλύτερους ε, γεωκτήμονες και, ε, και την ανησυχία του γιατί οι μεγάλοι καλλιεργητές ε, καρπώνονται τα, τα περισσότερα κονδύλια. Αυτή είναι η κρατούσα εντύπωση του ΕΛΚ, ότι πηγαίνουν ε, τα κονδύλια στους μεγάλους καλλιεργητές, ενώ αυτό δεν ισχύει, γιατί είναι δύσκολο ε, να λέει από τη μια ότι μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, αφιερώνεται στη γεωργία και τελικά καταλήγουν στις τσέπες των πολυεκατομμυριούχων. Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσουμε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν βρίσκω επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. Ο κύριο Άγνιου, διαδικαστικό, για αυτά που είπε ο Λουκ Φλάναγκαν. Ξέρω ότι η βασίλισσά μας δεν είναι ε, βασίλισσα της, και της Ιρλανδίας, αλλά δεν είναι μόνο βασίλισσα της Αγγλίας, είναι η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και φαντάζομαι θα με ευχαριστήσει η βασίλισσα ε, που το υπενθύμησα ότι δεν είναι μόνο βασίλισσα της Αγγλίας, αλλά του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm. Η κυρία Μπόσμαν θα μας εξηγήσει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενδιαφέροντα τα όσα άκουσα για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Ευπρόσδεκτο το ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος μειώνεται. Και όπως είπε η κυρία Κάλενμπαχ, το ποσοστό σφάλματος που διαπίστωσε το ελεκτικό συνέδριο ταιριάζει λίγο πολύ με την έκθεση ετησίων δραστηριοτήτων της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας. 2,02% είναι το ποσοστό σφάλματος το γενικό. Όπως είπε και το ελεκτικό συνέδριο, συμφωνεί. Μπορεί να το αντιστρέψουμε και να πούμε. Συνεπάγεται και αντιστρόφως ότι πάνω από 97% του γεωργικού προπολογισμού ξοδεύεται σωστά μιλάμε για ποσοστό σφάλματο, να μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχουμε τη βεβαιότητα για το που πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτό μπορεί και από, το σχεδιο γνωμοδοτησεω γνωμοδοτήσεως. Ένα-δύο σχόλια. Αναφερθήκατε κάνα δύο από εσά στη μεταρρύθμιση. 2015 ήταν το πρώτο έτος της μεταρρύθμισης. Σωστό αυτό. Πράγματι. Πρώτη φορά που εφαρμόσαμε τη μεταρρύθμιση των άμεσων πληρωμών. Όμως οι πληρωμές για το πρώτο έτος της μεταρρύθμισης έγιναν για το οικονομικό έτος 2016, πραγματοποιήθηκαν το 2016 στο ποσοστό σφάλματος δεν θα δείτε ε, το πώς επηρέασε μεταρρύθμιση των άμεσων πληρωμών αυτό. Ο κ. Μπέντας αναφέρθηκε στα αποκοπή, κατά αποκοπή ποσά και το απλουστευμένο κόστος για το 2016. Είχαν περιορισμένη δαπάνη στο νέο, ε, στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οπότε θα δούμε ότι θα συνεχιστεί η μείωση του ποσοστού σφάλματος στο δεύτερο πυλώνα. Επίσης, ευχαριστώ την κυρία Κάλεμπαχ που ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού τελικά ε, ε, κάνει σφάλμα. Μιλάμε για εντοπισμό αγροτεμαχίων και όχι εντοπισμό αγροτεμαχίων για χωματερές. Η λέξη χωματερή δεν ξέρω από πού προήλθε. Ήταν στην ΕΚΣ Επιτροπή Ελέγχου Υπολογισμού την τελευταία τετραετία και προσπαθούμε να αφαιρέσουμε αυτή την αναφορά. Ζητούμε βοήθεια, θα το εκτιμούσαμε. Για το σχέδιο έκθεση. Κανεί δεν το ανέφερε το σημείο 9. Εκεί γίνεται λόγο για το σύστημα εντοπισμού αγροτεμαχίων, το ΕΛΠΙΣ. Αναπόφευκτα θα υπάρχει αύξηση ποσοστού σφαλμάτων τα πρώτα χρόνια, αναφέρει, λόγω του συστήματο εντοπισμού αγροτεμαχίων του Δεν νομίζω ότι ισχύει. Το συστήσαμε το, από την αρχή, από το Άγιαξ, από το 97 χρησιμοποιούμε το σύστημα εντοπισμού μαχείο. Υπήρχε σφάλμα στο σύστημα εντοπισμού, αλλά δεν θα πρέπει να αυξηθεί λόγω της μεταρρύθμισης. Και το ελεγχτικό συνέδριο δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Όπως είπα, η έκθεση δεν αφορά τις μεταρρυθμισμένες άμεσες πληρωμές ακόμα. Κάποιοι αναφερθήκαν στο σημείο 4 για τις λανθασμένες, τις λανθασμένες αναφορές των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιτρόπου Χόκαν είπε ότι δεν πιστεύουν ότι στέλνουν λανθασμένα στοιχεία για τα σφάλματα τα κράτη-μέλη. Απλώς αυτά που ανακαλύπτουν τα σφάλματα κοινοποιούν, αλλά δεν βρίσκουν πάντα όλα τα σφάλματα. Γι' αυτό όταν κάνουμε την έκθεση ετησίων δραστηριοτήτων και υπολογίζουμε το σφάλμα, αυξάνουμε το ποσοστό σφάλματος που δηλώνουν τα κράτη-μέλη. Δεν το κάνουν σκόπιμα, απλώς δεν εντοπίζουν τα κράτη-μέλη μέσω των συστημάτων τους όλα τα σφάλματα. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Κάθε χρόνο εξετάζουμε τις εκθέσεις που μας αποστέλλονται στα στατιστικά στοιχεία και δεν βρήκαμε κάποιες περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων Καμιά φορά το σύστημα των κρατών μελών δεν διαπιστώνει όλα τα σφάλματα Εξού και το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Εθνικό Συνέδριο σε σχέση με τα ελέγχου που ενεργούν τα κράτη-μέλη. Εφόσον μιλάμε γι' αυτό, όπω είπε και η κυρία Κάλεμπαχ, βασιζόμαστε επί των ελέγχων που διενεργούνται στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η βάση του συστήματο. Δεν ακολουθούμε άλλη σειρά. Τι γίνεται στα κράτη-μέλη εξετάζουμε πρώτα. Μετά ρίχνουμε μια ματιά στους ελέγχους των κρατών μελών και βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό είναι το πλαίσιο των ελέγχων. Ευχαριστούμε για την γνωμοδότηση. Η έκθεση αναγνωρίζει ευτυχώς και είναι θετικό αυτό τη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβασή της. Ο κύριος Άγνιου για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρε, Ρώτησα ποιοι είναι οι κανόνε για τη συνεδρία των Επιτροπών στο Στρασβούργο. Απάντηση. Ούκα έλαβαν. Ευχαριστώ. Η απάντηση είναι ότι πράγματι, πράγματι, οι κανόνες του Προεδρείου προβλέπουν ότι συναντήσει συνεδριάσει συνεδριάσεις οδών κανονικών δεν πρέπει να διοργανώνονται στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια τη Συνόδου της αλλά είναι ρουτίνα οι παρεκκλήσεις που ζητούνται και χορηγούνται οι παρεκκλήσεις, εγκρίνονται. Άρα, κατ' εκτίμηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου διενεργούνται συνεδριάσεις αυτές. Εξετάζονται εξαιρέσει για τη διοργάνωση συνεδριάς των σκιωδών στο Στασβούργο. Γίνεται μια εκτίμηση τότε κατά πώ συνεδρίε των σκιωδών δημιουργεί προβλήματα για σημαντικές συναντήσεις ε, και εκδηλώσεις της Ολομελίας. Να μην συμπίπτουν ε, με ψηφοφορίες περίπτωση. Και είναι θέμα ερμηνείας των κανόνων. Αν δεν υπάρχει βασικός λόγος για απόρριψη, κανονικά προβλέπεται εξαίρεση και πραγματοποιούν συναντήσεις. Καταρχήν, έχετε δίκιο. Καταρχήν δεν προβλέπεται τέτοια συνάντηση. Άρα απαιτείται εξαίρεση. Πρέπει να ζητήσει κανεί εξαίρεση για να πραγματοποιηθούν αυτέ οι συναντήσει. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Νόησο. Έχω άλλη μια ερώτηση. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς υπολογίζεται το ποσοστό σφάλματος με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με ε, αναποσοστά 10, αναποσά 10.000 ευρώ. Πώς, πώς το υπολογίζεται αυτό παρακαλώ. Σας δίνουμε το λόγο και μετά θα δώσουμε στον κύριο Ιάχ το λόγο. Βεβαίως, εδώ μιλούμε για σφάλματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Τι μπορώ να σας πω εγώ όμως για μας. Το Συμβουλίο παίρνει ένα ε, δείγμα, αν θέλετε, για τον ε, πρώτο πυλώνα, μετά για την ε, ανάπτυξη της υπένθρου παίρνουν άλλες δαπάνες από τον τίτλο 2 του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν δείγματα τα οποία καλύπτουν τα κράτη-μέλη όχι αναπρόγραμμα και τελικά φτάνουμε για το IGF με ένα ποσοστό σφάλματος και μετά στο 2 για ε, τα ε, ανάπτυξη της με ένα άλλο ποσοστό σφάλματος. Στις αιτήσει δραστηριότητες στην έκθεση θα δείτε ότι το κάνουμε αυτό και για τις ε, άμεσες πληρωμές και για όλες τις ε, ε, δραστηριότητες τις οποίες έχουμε χωριστά. Εμείς λοιπόν βασιζόμαστε στα προγράμματα τα οποία στα αιτήσεις, αιτήσια, σε εκθέσεις που μας στέλνουν οι υπηρεσίες στατιστικής της κάθε χώρας και υπάρχει και οικονομική αξιολόγηση. Θα ήθελα τώρα να μου διευκρινίσετε το εξής. Το κύριο θέμα για μένα είναι όλα αυτά γίνονται βάσει προγραμμάτων, βάση ειδικών ποσών. Δεν είμαι η μόνη που θέτει τέτοιο πρόβλημα. Εάν είναι διαφορετική η κατάσταση, πολύ διαφορετική αν καταλαβαίνω καλά από αυτή που πιστεύουμε εμείς, μίλαμε πορτοκάλια, με... συγκρίνεται. Πρέπει να πω ότι συζητήθηκε για την μέθοδο που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο εκτενέστατο το θέμα. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Κένμπαχ, το ποσοστό σφάλματος τελικά πρέπει να πω ότι είναι παρεμφερές. Πρώτα απ' όλα για τις ε, αιτήσει. δραστηριότητες ήταν για το ΦΕΝΤΕΡ για την Κομισιόν 4,9 και 4,97 για τον ε, άλλο πυλώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για το ΦΕΝΤΕΡ. Απεφάσισε το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει τους ελέγχους στην Ευρώπη ε, διαφορετικά από ό,τι το έκαναν με τα κρατη Αλλά τελικά παρά το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικά δείγματα αν θέλετε κατέληξαν στο περίπου ίδιο ε, ποσοστό σφάλματος, γύρω στο 4,9%. Ο κύριος Φλάνναγκαν πάλι ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ένα από τα προβλήματα που βλέπω σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων με το ποσοστό σφάλματος είναι. Ξεκινάει μια κατάσταση από τις Βρυξέλλες, πάει στην φτάνει στους αγρότες. Για να μπορέσει κάποιος να έχει επιλέξιμο ε, αγροτική εκμετάλλευση, Πρέπει να πλήρει κάποια κτηρητήρια. Λένε όμως, κυρίως οι κτηνοτρόφοι, ότι ε, τα ζώα τους καταναλώνουν κάποιες ε, και επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο. Διαφωνούν όμως οι Βρυξέλλες. Η επιλεξιμότητα λοιπόν είναι κάτι το πολύ διαφορετικό για κάποιους. Λέει κάποιος στους αγρότες ότι κάτι που κάνουν για πάρα πολλά χρόνια δεν είναι σωστό, δεν είναι επιλέξιμη. Η Κομισιόν λέει κάτι διαφορετικό. Κάπου λοιπόν υπάρχει κάποιο σφάλμα. Είναι σφάλμα το ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί για τα, ε, για κοπάδια του κάποιες σκιές δωροτροφές, δεν είναι επιλέξιμο για κάτι, λέει η Κομισιόν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το παράδοξο, δηλαδή τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Κύριε Γιάρ, ας ολοκληρώσουμε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Για τη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών θα φροντίσουμε ε, με εκνευρίζει αυτή η συζήτηση γιατί είμαστε ενήλικες και μπορούμε να συνεδριάζουμε όποτε θέλουμε και όποτε θέλουμε οι σκιώδεις συγγητές. Ε, ανέκαθεν είχα πει ότι με, μου την έδινε αυτό το θέμα. Με εκνεύριζαν οι περιορισμοί αυτοί καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας να μην μπορούμε να συνεδριάζουμε όπου, θέλουμε. Και για την πρώτη συνεδρίαση δεν ζήτησα εγώ τίποτα. Έγινε τέλος πάντων, ότι έγινε έγινε, τα παθήματα μαθήματα, αλλά νομίζω ότι είμαι ελεύθερος να έχω συναντήσει με όποιον θέλω, είμαι ελεύθερος να έχω επαφές με τους συναδέλφους. Εντάξει, σέβομαι τους κανόνες, αλλά κανένας ε, δεν μου είχε πει ότι διαφωνεί με τη διοργάνωση της ε, συνεδρίας του για τον και παρόλα αυτά τελικά δεν έγινε, γι' αυτό και εκνευρίστηκα. Τώρα, για το ποσοστό σφάλματος. Ε, το σφάλμα δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο ή απόλυτο. Αποφασίσαμε ότι θα χρησιμοποιούμε δείγματα, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και αυτό θα καθορίζει το ποσοστό σφάλματος. Και το ποσοστό σφάλματος δεν δείχνει το εύρος των οικονομικών ζημιών. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι 3% είναι ένα γενικό ποσοστό σφάλματος που αντιπροσωπεύει χ δισεκατομμύρια ευρώ και το τάδε πρόβλημα στον ε, προϋπολογισμό. Το ποστό σφάλματος δεν λέει τίποτα για τις οικονομικές ζημίες. Και το λέει αυτό και ο εισηγητής της κύριας έκθεσης. Είπε ότι λαμβάνουμε τα τελικά ποσά και με το ποσοστό σφάλματος καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι σωστό πάντα αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι διαφορετικά τα σφάλματα και μερικές φορές ε, δεν έχουν όλα τα σφάλματα τις ίδιες ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Και ε, το 2,2 είναι αρκετά αξιοπρεπές ποσοστό τελικά. Μπορούμε να λέμε και να μιλάμε ώρες ολόκληρες για το ποσοστό σφάλματος. Τώρα, το ποσοστό σφάλματος στον πρώτο πυλώνα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό του δεύτερου πυλώνα. Και πολλά εξαρτάται και από τους αποδέκτες, από τους δικαιούχους. Και οι γεωργοί που εμπίπτουν στο πρόγραμμα άμεσων ενισχύσεων δίνουν μάχη κάθε χρόνο ε, και χρειάζεται να υποβάλλουν τι αιτήσει του στη διοίκηση και γίνεται ένα είδο αμοιβαία κατάρτιση Στις, σε μερικέ ε, αγροτικέ ζώνες, μερικοί γεωργοί μια φορά ε, μόνο στη ζωή τους κάνουν ε, αυτές τις αιτήσει. Και αυτό είναι πιο, είναι πιο εύκολο να κάνουν λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Υπάρχουν πιο πεπειραμένοι γεωργοί που έχουν υποβάλει πολλές φορές παρόμοιες αιτήσει και Άλλοι που ανανεώνουν τις γεωργικές τους εκτάσεις μπορούν να το κάνουν μια φορά μόνο στη ζωή τους. Γι' αυτό και ίσως σε τέτοιες περιπτώσεις το ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο. Και θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των ποσοστών σφαλμάτων, γιατί ίσως εκεί έχουμε φαινόμενα διαφθοράς. Πάντως, ε, συνήθω μιλούμε για γεωργούς που μια στις τόσες, μια ε, πολύ σπάνια υποβάλλουν τέτοιες αιτήσει. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε ή να παραβελούμε το δεύτερο πυλώνα μόνο και μόνο επειδή έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις γι' αυτόν. Τώρα, για τα νέα προγράμματα και την ανάγκη να αποφύγουμε γραφειοκρατικές ε, διατυπώσεις, εμείς θέλουμε να ε, στηρίξουμε επενδυτικά προγράμματα ιδιαίτερα στις αγροτικές ζώνες και να μπορούν να υποφελούνται οι γεωργοί από αυτά τα προγράμματα. Όταν έχουμε όμως κανονισμούς και κανόνες θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και να, μην, και να είναι ε, συμβατοί μεταξύ τους οι κανονισμοί, όχι αντιφατικοί, περιπλέκοντας έτσι τη γραφειοκρατία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Επίσης διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά μικρή εμβέλεια προγράμματα από διάφορα επενδυτικά ταμεία, αλλά το βασικό είναι να αποφευθούμε ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Θέλουμε τα προγράμματά μας ε, να έχουν αποτελέσματα στην Ήπεθρο, στις αγροτικές ζώνες. Και σίγουρα η ενίσχυση της γραφειοκρατίας ε, δεν είναι προς όφελος των προγραμμάτων, ούτε προς όφελος των γεωργών που θα είναι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων. Και προσοχή, μπορούμε να μιλούμε για τους στόχους μας, μπορούμε να μιλούμε για τη λειτουργία της ε, ευρωπαϊκής Ιωρικής πολιτικής, μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες για τα θέματα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τις μεμονωμένες αποφάσεις που λαμβάνονται. Και η εφαρμογή των αποφάσεων δεν μπορεί να είναι καλύτερη από τις χρήσεις αποφάσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπερφορτώσουμε την έκθεση με λεπτομέρειες, με τι μας δυσαρεστεί. Γιατί θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άμα από εσά εξαρτάται σε τελική ανάλυση η λήψη της απόφασης. Η δική σας απόφαση δεν ήταν άρτια. Ε, εμείς απλώς την ε, εκτελούμε. Δεν φταίμε αν η απόφαση η ίδια ήταν κακή. Ελπίζω να σας απάντησα στις απορίες. Θα γίνει και άλλη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών πριν καταλήξουμε σε συμφωνία. Πάντως γενικώ θεωρώ ότι είχαμε θετικά μηνύματα από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της γεωργίας γιατί δεν έχει αυξηθεί το ποσοστό σφάλματος και γενικώ οι χρήστες ε, του προπολογισμού της γεωργίας χαίρουν συγχαρητηρίων γιατί χρησιμοποιούν καλά τα κονδύλια και με χαμηλό ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Να σας υπενθυμίσω την 5η Δεκεμβρίου το μεσημέρι που λύγει η προθεσμία της κατάθεσης των τροπολογιών. Περνάμε τώρα στο τελευταίο πρωινό σημείο της ημερήσιας διάταξη. την παρουσίαση της γνωμοδότησης της κυρίας Ούλρη και Νταντσίλα για τις συνθήκε εργασία και την επισφαλή απασχόληση. Δυστυχώ η κυρία Νταντσίλα απουσιάζει. Άφησε στο πόδι της όμως τον κύριο Ντεκάστρο που θα μας παρουσιάσει την ε, γνωμοδότηση της κυρίας ε, Νταντσίλα θα εγκύψουμε στην ιδιαίτερη κατάσταση της γεωργίας και στην επισφάλεια των θέσεων απασχόλησης ε, στον κλάδο αυτό. Κάτι που βιώνουμε όλοι μας και στις πατρίδες μας. Και να υπενθυμίσω και πάλι την διορία για την κατάθεση των τροπολογιών. 5 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, λίγη προθεσμία. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Δεκάστρο για να μας παρουσιάσει την αγνομοδότηση της κυρίας Νταντσίλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γιώργικα για τη δουλειά που έκανε και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα εδώ. Αυτή η γνωμοδότηση προορίζεται προς την Επιτροπή Απασχόλησης και επικεντρώνει προσοχή της επί των επισφαλών συνθήκων εργασίας που αφορά τους γεωργούς και τους ασχολούνται με το αγροτικό τομέα ε, που είναι, εκτίθεται πιο πολύ σε αυτόν τον κίνδυνο από τι άλλε τομεί. Υπογραμμίζει ότι ο γερικό τομέα υπόκειται σε διάφορου εξωτερικού παράγοντε αλλαγή των τιμών και των αγορών, αλλαγή του κλίματο και έτσι είναι αβέβαιη η δυνατότητα απασχόληση. Η Επιτροπή, Επιτροπή και τα κάτι μέλη ε, θα πρέπει να προωθήσουν διάφορα εργαλεία για να στηρίξουν το εισόδημα και να εφαρμόσουν και τα φυστάμενα μέσα όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει ότι αυτό είναι αναγκαίο αναλύοντας την περίπτωση των εποχιακών εργαζομένων για τους οποίους ζητά την αναγνώριση ενός νομικού καθεστώτος για αυτούς ούτως ώστε να μπορούν να εγγυηθούν σε αυτούς προστασία κοινωνική. Απαιτεί λοιπόν την προσοχή στην ειδική περίπτωση των εποχιακών εργαζομένων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κατάσταση επισφαλών συνθήκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μελη καλούνται να ρυθμίσουν τη θέση, την κοινωνική και νομική αυτών των ανθρώπων και να τους παράσχει κοινωνική προστασία. Η συγγήτρια ε, λαμβάνει υπόψη ότι οι νέοι και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να βρουν εργασία στην Ήπεθρο και να ξεκινήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Μία υποστήριξη ειδική θα πρέπει λοιπόν να προβλέπεται και για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων. Γι' αυτό το Ταμείο για τους Νέους Γεωργούς και τα προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις, στην Ήπεθρο θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν μια απασχόληση ποιοτική ε, με τη σωστή αμοιβή. Υπογραμμίζεται τέλος ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των διάφορων φορέων προνοίας στην Ήπεθρο για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας και για την ενίσχυση της ασφαλείας και της ευημερίας στον τόπο εργασίας για να διευκολυνθεί έτσι η ένταξη όλων των κατηγοριών των εργαζομένων στο γεωρικό τομέα, των νέων και των γυναικών συμπεριλαμβανομένων και πιο συγκεκριμένα να λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση των εποχιακών εργαζομένων. Ευχαριστώ και προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 5 Δεκεμβρίου του 2016 στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Δικάστρο για τις διευκρινήσεις. Η κυρία Σέντρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, το θέμα αυτό των επισφαλών συνθήκων εργασία στην θα ήθελα τώρα να τονίσω το εξή. Εκτό από τι ε, συνθήκε που αφορούν τους μισθωτού και τους εργαζόμενους και τι εργαζόμενου τους εποχιακού, οι συνθήκες που επιβάλλει η ΚΑΠ που όλο και περισσότερο οδηγεί σε τιμές και εισοδήματα χαμηλότερα για όλους τους αγρότες είναι κάτι το οποίο κάνει την εργασία όλων όσων απασχολούνται στην τομέα πιο επισχαλή, πιο πρόσκαιρη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι προβλέπω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες για να μπορέσω να εμπλουτίσω αν θέλετε περισσότερο και με το θέμα αυτό την έκθεση. Σας ευχαριστώ. κύριε Ριμπέρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εργασία που έγινε από την συνάδελφο και να πω το εξή. Πιστεύουμε ότι κάποια θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση να τα παρουσιάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειε. Θα τονίσουμε όπω και ο κύριος Δεκάστρο, οι πρόσχερε συνθήκε εργασία έχουν να κάνουν και με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, με τι εμπορικέ πρακτικέ και με τα θέματα της ε, διανομής που υπάρχουν στην ε, τομέα αυτό των αγροδιατροφικών και κυρίως ε, έχουν να κάνουν και με θέματα πιο έντονα και με προβλήματα πιο έντεκα για τις υπερπεριφερειακές επιτροπές τις οποίες υπάρχουν όλο και περισσότερο τέτοιου είδους κακές συνθήκες. Εμείς θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι στα διάφορα κέντρα αγροτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να δίδονται ε, διαφορετικές απαντήσεις στα θέματα που τίθενται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν κάποιες συνθήκες να τυποποιηθούν ώστε να ισχύουν ήδη κανόνες παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες θα πρέπει κυρίως να είμαστε υπέρ των ε, ελάχιστων ε, ε, θετικών συνθήκων που δίνουν του εργαζόμενου, όπω το θέμα της κατάρτισης, το θέμα του συνδικαλισμού. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταπολεμήσουμε την μη δεδηλωμένη εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μηχανισμούς για να ε, συντονιστούμε με τον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα που ε, ορίζει τις συνθήκες εργασίας στον τομέα αυτό ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σωστές προτάσεις, να συντονιστούν οι διάφοροι τομείς, ώστε οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας να είναι στο ελάχιστο δυνατό ποσοστό. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα ήταν ε, ενδιαφέρον να ζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία μέγα εκστρατεία ενημέρωσης των εργαζόμενων και των ε, φορέων που απασχολούν αυτού του τύπου εργατικό δυναμικό ώστε να μην ισχύουν πλέον πρόσκαιρες συνθήκες εργασίας και επισφαλής και να μπορέσουν να ενημερωθούν σωστά οι εργαζόμενοι ώστε να μην είναι αντικείμενο καταχρήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω η συγγητρία και θα πρέπει να σας πω και στη δική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή Πασχόλησης ασχολούμαι με αυτό το θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και με τη συνεργασία όλων πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chair. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Οι συνθήκες εργασίας στην Ήπεθρο είναι δύσκολες, επισφαλείς και επικίνδυνες. Η γεωργία εξαρτάται κατά πολύ από τους πιο ευάλωτους εργαζομένους, όπως εποχιακούς εργαζομένους, μετανάστες και καμιά φορά οι συχνάς, ε, οι οποίοι δεν έχουν καν τα σωστά έγγραφα. Οι γεωργοί λοιπόν, οι εργαζόμενοι στη γεωργία δουλεύουν πολλές ώρες, βγάζουν λίγα και είναι ασταθής η εργασία τους. Η γεωργία είναι επικίνδυνη η απασχόληση. Έχει κανεί κίνδυνο να τραυματιστεί. Και έχουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό θανατηφόρων τυχημάτων. Η απασχόληση στη Γεωργία σήμερα αλλάζει διαθροτικά. Και είναι πολύ πιο σπάνιο να μόνιμη απασχόληση στη Γεωργία. Εξαρτάται η Γεωργία σε μεγάλο βαθμό από χειρονακτική εργασία, περισσότερο από άλλου τομεί. Και αυξάνεται το θηλυκό εργατικό δυναμικό, πρόσδεκτο σχόλια για το κείμενο. Για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Εποχιακή εργασία. Είναι κοινή στην ευρωπαϊκή εργασία, είναι δομικό στοιχείο του τομέα. Αυξάζεται η δαπάνη της σταθερής εργασίας στο κόστος της. Γι' αυτό επιτυχώς έχουμε εφαρμόσει προγράμματα για να δίνουμε μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια απασχόληση εποχιακούς εργαζομένους. δεν θα πρέπει να υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα μέσω των συμβάσεων ίσως. Θεωρείται ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα δεν έχουν πολλά προσόντα, οπότε τίθεται και θέμα ε, επαγγελματικής κατάρτισης για να βελτιωθεί η θέση τους. Προσφέρει η Γεωργία κάποιες θέσεις εργασίας που απαιτεί μεγάλα προσόντα, αλλά δεν υπάρχει σωστή εικόνα για τις ανάγκες οι γεωργοί μπορεί να συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση του ε, πληθυσμού. Έχουμε πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε τη μίση του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Αλλάζει η γεωργία, μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις επασχόλησης. Άρα πρέπει να εστιαστούμε επίσης επί μισθωτής γεωργικής εργασίας. Πρέπει να αποφύγουμε τη μετάλλευση των μεταναστών στη γεωργία από διάφορους επιτίδιους σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης και στη Σουηδία. Εργαζόμαστε η Γεωργία είναι από την Υποσαχάρια Αφρική, από την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και ε, ε, εργάζονται για πενιχρές αμοιβέ, υπό άθλες συνθήκες και, στα, και κοιμούνται κοντά στα θερμοκήπια, στα αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Μέχρι και 5 ευρώ την ημέρα μπορεί να βγάζουν για 10-12 ώρες εργασίας. Πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό. Είναι μια μάστιγα. Δεν θα ενταχθούν οι πρόσφυγες αν δεν δείξουμε κάποια αλληλεγγύη προς αυτούς. Ευχαριστώ τους συγγητές για την καλή δουλειά που έκαναν και θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Ούτως ώστε οι τροπολογίες που θα υποβάλουμε να αντικατοπτρίζουν τις πρώτερες ε, παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Ο κ. Φλάναγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την έκθεση. Δυστυχώς, κανονικά όταν μιλάμε για επισφαλή εργασία και συνθήκες εργασίας, μιλάμε για τη μειοψηφία. Όμως τη Γεωργία, με την κρίση που αντιμετωπίζει, μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία, τεράστια πλειοψηφία. Αν επισφαλής απασχόληση και συνθήκες εργασίας σημαίνουν να παίρνεις λιγότερο το προϊόν από ό,τι σου κοστίζει να το παράγεις, αυτό καλύπτει όλους σχεδόν. Υπάρχουν και άνθρωποι σε πιο επισφαλείς θέσεις, άμα δεν είναι διοκτήτης της γης και είναι εποχιακός εργαζόμενος. Άρα πρέπει να προστατευτείς. Ο πρώτος τρόπος να τους προστατεύσεις, ο πιο σημαντικός, όπως είπα και πριν, για τη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ή τη βασίλισσα της Αγγλίας που εμίλησα. Λοιπόν, πηγαίνετε σε ένα πάθη γενεθλίων. Αν ένα παιδί φάει όλο το, την τούρτα δεν θα φάνε τίποτα τα άλλα παιδιά. Γι' αυτό είναι τόσο επισφαλής η κατάσταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα σας. Όταν έγινε διαπραγμάτευση για την κοινή αγροτική πολιτική ήμουνα καινούριο και σκέφτηκα. Πώς μια οργάνωση γεωργών μπορεί επιτυχώ να πείσει τα μέλη τη ότι η πλειοψηφία θα τα κατάφερε καλύτερα με λιγότερα χρήματα. Το κατάφεραν. Του κατάφεραν να κάνουν πορεία προ την ποτέ να διαμαρτυρηθούν ο, για κατά ποιο δίκαιης ε, κατανομής μέσω της ΚΑΠ. Το υπαριθμό να έπρεπε να κάνουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ΚΑΠ θα εφαρμοστεί σωστά και στη χώρα μου. Δεν εφαρμόζεται σωστά και σε άλλες χώρες, ναι. Δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε αυτό. Διότι έχουμε ισχυρέ δυνάμεις που μάχονται εκείνους που δεν έχουν πάρα πολλές ε, δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μπαρέρο Φλόρες. Ποια είναι η θέση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συζητήσεις επί της εκθέσεως. Μας ενδιαφέρει το θέμα της επισφαλούς απασχόλησης και ο πρόεδρος Γιουγκέρα από την αρχή μίλησε για τα 3α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την κοινωνική Ευρώπη και για τον κοινωνικό πυλώνα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας για το συγκεκριμένο αυτό θέμα της επισφάλειας της απασχόλησης και τη δική σας έκθεση θα την προσέξουμε ιδιαίτερως και την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ κύριο Στεκάστρο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις της σημειώνω και θα ενημερώσω την ε, Γιώργη Καντάντσιλα και ευχαριστώ για τις τροπολογίες και για τη συνεργασία που... Α, και των προτέρων για τη συνεργασία με τους συναδέλφους και τις τροπολογίες που θα υποβάλουν. Ευχαριστώ. Προθεσμία τροπολογία είναι 5 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεισφορά σας και θα είναι πολλές τροπολογίες, δεν αμφιβάλλω, διότι είναι μεγάλο το διακύβευμα. Πολύ σημαντικό. Κερδίσαμε χρόνο. Θα δώσω το, το λόγο στον πραγματικό πρόεδρο, τον κ. Σικέρσκι. Θα του δώσω το σφυράκι που κατέφθασε και συνεδρίσει των συντονιστών στις 11 και 4 θα γίνει αντί στις 11 και μισή. Ήδη σας ενημερώσαμε. Θα τα ξαναπούμε και το απόγευμα στις 3 θα είδατε ότι το ραντεβού είναι στην αίθουσα του εμικυκλίου, στο εμικύκλιο, όπου θα συνεδριάσει η Επιτροπή το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο πρωινό και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια των εργασιών.